θα αρχίσει να τρέχει από αύριο 20 Φεβρουαρίου του 2009. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο για έγκριση στην αρχή της επόμενης συνόδου και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις θα προωθήσω τα ψηφίσματα που υιοθετήσαμε στα πρακτικά αυτά.